περίοδου Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διακοπή στις 24 Μαΐου του 2012. Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 24 Μαΐου του 2012 είναι στη θέσή σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις στα πρακτικά. Όχι και ως εκ τούτου εγκρίνονται. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ε, χαιρετήσω